αφορά τον κύριο Έντουαρντ Ραούλ Χελβίκ που υπέβαλε την ε, παρέτησή του από την εντολή του ως Ευρωβουλευτή με ισχύ από τις 2 Μαρτίου 2015 και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφη 1 και 3 του κανονισμού το, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την, ε, ε, την